Λοιπόν, αγαπητοί μου συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Έχουμε ένα εργαστήριο με θέμα την εξέλιξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε κράτη-μέλη που υπάγονται σε προγράμματα της Τρόικας και κράτη-μέλη που έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή των προγραμμάτων και έχουν βγει από τα μνημόνια δηλαδή. Καλώς ορίζω και ευχαριστώ θερμά ε, το ε, θεματικό τμήμα Α το οποίο παρακαλέσαμε να ε, έρθει για ένα τέτοιο εργαστήριο. Καλώς ορίζω τους διάφορους εμπειρογνώμονες που έχουμε σήμερα στην ημερασία διάταξη. Ο Ρικάρτο Ροτρίγκης Κοντρέρα, είναι ο πρώτος από το Eurofound, η Μαρία Λαπά Κάμπο Λίμα από το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, η Αουρόρα Τρίφ από το Πανεπιστήμιο της Πόλη του Δουβλίνου ο Πίτερ Ρίγνη από το ελλαδικό Κόγκρεσο ε, και την αριστεία Κουκιαδάκη και ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Ε, τα ονόματα τα ελληνικά κυρίως με δυσκολεύουν πολλές φορές. Ε, ε χαίρομαι που ήρθατε να συζητήσουμε. Έχουμε 45 λεπτά τώρα μόλις μέχρι το πρώτο διάλειμμα για το γεύμα και θα συνεχίσουμε στις 3.30. Ε, με τη δεύτερη ενότητα. Να πω δύο λόγια ε, για το υπόβαθρο και το ιστορικό. Γιατί ασχολήθηκε η Επιτροπή μας με το θέμα αυτό. Καταρχάς πρέπει να πω ότι έχουμε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2014 το οποίο ασχολήθηκε με τα θέματα απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές ε, στα πλαισία των προγραμμάτων της Τρόικας και στη δική μας Επιτροπή έχουμε μια ομάδα παρακολούθησης για τα νέα δικαιώματα, τα εργασιακά και τα κοινωνικά στην Ελλάδα. Μας παρακάλεσε η ελληνική κυβέρνηση να δραστηριοποιηθούμε και ένα τρίτο θέμα που μας απασχολεί και θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει που είναι ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει κάπως να αναζωογονηθεί, για να το πω έτσι, να αφυπνιστεί, το λέω πολύ προσεκτικά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν κάνουμε τη σημερινή μας ακρόαση και χωρίς περαιτέρω εισαγωγή θα ήθελα να δώσω μέσω το λόγο στον Ριτρά, ε, Ρικάρδο Ροντρίγκες Κοντρέρα στη Eurofound για να μας κάνει την παρουσίασή του για 10 λεπτά ή δυνατόν. The microphone. το Microphone. Yes, it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair, again. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω μία πρόσφατη μελέτη μας, μία μελέτη της Eurofound, όσον αφορά την εξέλιξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Καλύψαμε μία μεγάλη χρονική περίοδο Θεωρούμε ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν συμβεί στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια, τουλάχιστον από το τέλος της δεκαετίας του 1990. Κάναμε λοιπόν μία προσπάθεια να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης και να δούμε τελικά πώς εξελίχθηκε στο χρονικό αυτό διάστημα το όλο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θεωρήσαμε ότι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου να αξιολογήσουμε τις λογικές διαπραγματεύσεις και να δούμε πώς αυτές διαμορφώνονται στην ε, Ευρώπη. Η βασική ιδέα εδώ πέρα ήταν να κάνουμε μια χαρτογράφηση των ε, τρόπων που ρυθμίζονται και των τρόπων που διεξάγονται λογικές διαπραγματεύσεις, όπως σας είπα, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα. Αληθεύει, όπως θα το δούμε και λίγο παρακάτω, ότι έχουν γίνει πολλές έρευνες και μελέτες τα τελευταία χρόνια, ιδίω στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, για το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αρχίζουν σιγά σιγά και αναδύονται κάποιες τάσεις. Άλλες πάλι είναι πιο μακροχρόνιες τάσεις και ξεκίνησαν και πριν από την εμφάνιση οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι λοιπόν η βασική ιδέα που διέπει την ε, μελέτη αυτή, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε μάλιστα και από την ιστοσελίδα της Eurofound και έχω φέρει μαζί μου βέβαια και κάποια αντίγραφα. Η μελέτη αυτή ασχολείται μόνο με τις ε, εξελίξεις όσον αφορά τα κεντρικά στοιχεία των στοιχικών διαπραγματεύσεων. Δεν αφαιρόμαστε καθόλου σε μηχανισμούς καθορισμού των μισθών, δεν αναφερόμαστε στο χρόνο εργασίας και το ωράριο εργασίας ή σε άλλα επιμέρους ζητήματα. Για τα ζητήματα αυτά υπάρχουν και επιμέρους μελέτες της Eurofound. Εμείς αποφασίσαμε στη συγκεκριμένη μελέτη να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των εμπλεκομένων μερών, πώς διαμορφώνουν τις τουρκικές διαπραγματεύσεις, ποιο ρόλο επιδραματίζουν, ποια διαδικασία ακολουθούν, πώς εφαρμόζονται στη συνέχεια οι συλλογικές συμβάσεις που προκύπτουν από τις τουρκικές διαπραγματεύσεις και να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα, πόσες τέτοιες συμβάσεις και συμφωνίες έχουμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχουν στην πράξη. Η μελέτη αυτή ακολουθεί μια κλασική, θα έλεγα, συνήθι δομή. Βλέπουμε τους βασικούς παράγοντε τους βασικούς φορείς, τις βασικές διαδικασίες, και νομίζω ότι ε, μπορούμε μέσω της μελέτης αυτής να δούμε και όλη αυτή τη συζορευμένη εμπειρία και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει Eurofound τα τελευταία χρόνια. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε πολλές μελέτες και έρευνες, οι εκθέσεις τις οποίες έχουμε εκπονήσει και έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις και είναι μελέτες βέβαια ιδιαίτερα λεπτομερείς. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη μας ήδη την ε, μελέτη αυτή και όλες αυτές τις μελέτες για να καλύψουμε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Επίσης, ε, χρησιμοποιήσαμε υφιστάμενες ερευνητικές ε, μεθόδους, καθώς επίσης και την πανεπιστημιακή βιβλιογραφία και άλλες πηγές, προκειμένου να καταφέρουμε να εμπλουτίσουμε τη μελέτη αυτή και βέβαια και τις πληροφορίες μας δώσαν οι ανταποκριτές μας, οι απεσταλμένοι μας, στα κράτη-μέλη. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τους ε, φορείς, τους παράγοντες αυτούς καθεαυτούς. Η πρώτη εξέλιξη που μας απασχόλησε ήταν πώς εξελίσσονται οι ίδιοι οι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και αναφέρομαι σε εκπροσώπους εργαζομένων, εκπροσώπους εργοδοτών. Ποιο ήταν ο ρόλος τους τα τελευταία 15 χρόνια. Στη συνέχεια, και ενδεχομένω το ξέρετε αυτό, βλέπουμε ότι καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μια αξιολόγηση αυτής της κατάστασης. Ξέρω ότι πολλές φορές τα στοιχεία τα οποία έχουμε δεν είναι πλήρη αξιόπιστα. Γενικότερα πάντως είναι αποδεκτό το γεγονός ότι από τη μία πλευρά υπάρχει μια γενικότερη μείωση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ε, συμμετοχής σε αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, μειώνται δηλαδή τα μέλη τους και από την ε, άλλη πλευρά βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί περισσότερο από τη δεκαετία του 90 και μετά. Στο δεξιό τμήμα τη διαφάνειας, στην δεξιά γραφική παράσταση, βλέπετε τη μείωση τη συμμετοχής στις συνδικαλιστικές οργανώσεις από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα και βλέπετε ότι ε, η μείωση αυτή είναι γενικευμένη, μολονότι σε κάποιες ώρες έχουμε πιο σταθερά στατιστικά δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν μια αποκλίνουσα εξέλιξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ αντικειμενικά. Διαφέρει η κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη ή από τον οικονομικό κλάδο στον άλλο. Στην αριστερή γραφική παράσταση βλέπετε τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πάνω από 10 εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες έχουν μια κάποια μορφή συνδικαλιστική σύμβαση ή προβλέπουν τουλάχιστον συνδικαλιστικές διαπραγματεύσεις. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε λοιπόν ποιε είναι οι γενικότερε τάσει που αναδύονται αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχή των οργανώσεων κοινωνικών εταίρων στι λογικέ διαπραγματεύσει. Έχουμε τι οργανώσει εργοδοτών και τι συνδικαλιστικέ οργανώσει. Δεν υπάρχει εξέλιξη στις χώρες αυτές που βλέπετε πάνω αριστερά, αυτές που παρουσιάζουν σταθερότητα. Έπειτα βλέπετε μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ανατολικές και δυτικές χώρες. Χώρες οι οποίες έχουν μια μακροχρόνια παράδοση όσον αφορά τον εργασιακό κοινωνικό διάλογο και τις χώρες εκείνες της ε, Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης οι οποίες έχουν διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε επίσης πολύ σημαντική μείωση τόσο στις οργανώσεις εργοδοτών όσο και στις οργανώσεις ε, τις συνδικαλιστικές στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Και ουσιαστικά στη διαφάνεια αυτή βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα. Έχετε μια σφαιρική απεικόνηση τη κατάσταση όσον αφορά την, ε, τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων και το ποσοστό συμμετοχής σε αυτές και βλέπουμε ότι σε ορισμένες χώρες οι συλλογικές διαπραγματεύσεις επηρεάζονται από τον τρόπο που γίνεται ο κοινωνικός διάλογος, αν συμμετέχουν δηλαδή δύο ή τρεις φορείς, αν έχουμε διμερείς ή τριμερείς διαπραγματεύσεις. Εν γέννη, στην χρονική αυτή περίοδο που εξετάσαμε, ο κοινωνικός διάλογος είτε είναι τριμερή είτε είναι διμερή, εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό. Ιδίω στα πλαίσια τη πρόσφατη οικονομική κρίση. όπου είδαμε ότι ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση χρησιμοποίησαν τον κοινωνικό διάλογο ω αποτελεσματικό εργαλείο για να επιφέρουν αλλαγέ και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασία. Στην διαφάνεια αυτή βλέπετε το δεύτερο τμήμα των σημαντικότερων αυτών εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις λογικές διαπραγματεύσει και κυρίως με τη διαδικασία αυτή καθεαυτήν. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ίδια την έκθεσή μας. Εγώ προσπάθησα απλώς στη διαφάνεια αυτή να σας δείξω σχηματικά τις πιο σημαντικές εξελίξεις και είμαι πεπισμένο ότι οι συναδελφοί μου θα είναι σε θέση να σα δώσουν πολλέ περισσότερε λεπτομέρειε όσον αφορά για παράδειγμα τις αποκλήσεις παρουσιάζονται συλλογικέ συμβάσει. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο λεγόμενο μηχανισμό επέκταση, τη ισχύω, τη κάλυψης μια συλλογική σύμβαση. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στη δυνατότητα μεταβίβαση, μεταφορά ορισμένων πτυχών μια συλλογική σύμβαση σε άλλου οικονομικού κλάδου. Εν συντομία, θα λέγαμε ότι ε, έχει επιταχυνθεί πολύ σημαντικά αυτό το φαινόμενο της απόκλησης των συλλογικών συμβάσεων από αυτές που είχαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Από το 2008 και μετά, σε ορισμένες χώρες και κυρίως στις χώρες που αναλύουμε, για παράδειγμα Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ελλάδα, έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές και έχουν προβλεφθεί νέοι τρόποι συλλογικής διαπραγμάτευσης, οι νέες αποκλίνουσες πρακτικές ή ακόμα και η προσωρινή δυνατότητα να εγκαταληφθεί μια γενική συλλογική συμφωνία, διακλαδική για παράδειγμα. Βλέπετε λοιπόν ότι χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί μηχανισμοί σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά ιδίω σε ορισμένες χώρες, τις τέσσερις ανέφερα αλλά και σε άλλες όπως την Ισπανία, βλέπουμε ότι έχουν γίνει αυτή τη στιγμή ρυθμιστικές αλλαγές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αποκλίνει κανείς περισσότερο από την γενική διακλαδική συλλογική σύμβαση που ίσχυε στο παρελθόν απαρέκλητα. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε πάλι τις ε, βασικές αποκλίνουσες ε, διαδικασίες που ισχύουν τώρα σε ορισμένα κράτη-μέλη και όπως σας είπα ξεκίνησαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα. Το πρώτο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί εδώ πέρα είναι ο κεντρικός χαρακτήρας των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε ορισμένες χώρες που υπήρχε ένα παγιεμένο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα πράγματα δεν έχουν τροποποιηθεί. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην πράξη είναι ότι από το 2008 και μετά έχει αυξηθεί το φαινόμενο της αποκέντρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ιδίως σε κάποιες νότιες χώρες. Αυτή η διαδικασία αποκέντρωσης και γενικότερα όλες αυτές οι αποκλίνουσες διαδικασίες σε σχέση με το παγιωμένο παρελθοντικό μοντέλο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα ζητήματα συντονισμού. Τι λέμε όταν χρησιμοποιούμε τον όρο συντονισμό. θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς συντονίζονται αυτές οι συλλογικές συμβάσεις σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους κλάδους. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κλαδικές τέτοιες συλλογικές συμβάσεις ή μπορεί να έχουμε συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης μόνο. Ή μπορεί να υπάρχει συντονισμός ή να μην υπάρχει συντονισμός ανάμεσα σε συμβάσεις που συνάπτονται στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή ίδιος οικονομικός κλάδος ή ακόμα και ίδια επιχείρηση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αναλύσουμε εδώ πέρα το φαινόμενο του συντονισμού. Είδαμε ότι και αυτό μειώθηκε από το 2008 και μετά, ιδίως στις χώρες οι οποίες ακολουθούν ένα πρόγραμμα της Τρόικας, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα. Και σε έναν βαθμό έχει μειωθεί ο συντονισμός συλλογικών συμβάσεων και στην Πορτογαλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η αποκέντρωση πλέον αποτελεί παγιωμένη τάση. Είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν από την κρίση, αλλά είναι μια τάση που συνεχίζεται τώρα και μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα, και ολοκληρώνω, στη Γερμανία, για παράδειγμα, ή σε κάποιες βόρειες χώρες όπου έχουμε συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων, η τάση της αποκέντρωσης έχει γίνει με τρόπο πολύ συντονισμένο. Δηλαδή, έχουμε κοινωνικό διάλογο, συμμετέχουν οι οργανώσεις εργοδοτών και οργανώσεις εργαζομένων και καταφέρνουν από κοινού να συμφωνήσουν επί συγκεκριμένων κανόνων και να μην αποδυναμώσουν το τελικό αποτέλεσμα της συλλογική διαπραγμάτευσης. Και περνάω και στην τελευταία μου διαφάνεια, κύριε Πρόεδρε. Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι οι τάσεις αυτές που σας περιέγραψα και που αναλύονται πολύ περισσότερο στη μελέτη μας. Είναι τάσεις που ε, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης επηρεάζουν έναν τελικό δείκτη τελικά, ο δείκτης της κάλυψης της λογικής ε, σύμβασης. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πόρισμα της μελέτης μας. Στον πίνακα αυτό που έχετε ενώπιόν σα, βλέπετε ότι στα τέλη τη δεκαετία του 90 η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων ήταν τη τάξη του 68%. Σε σχέση δηλαδή με το σύνολο των εργαζομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτό μειώθηκε λίγο στη συνέχεια το 2007, λίγο πριν ξεκινήσει δηλαδή η οικονομική κρίση, φτάσαμε τότε το 66%. Αλλά από το 2008 και μετά, τα τελευταία δηλαδή αυτά χρόνια, το συνολικό ποσοστό κάλυψης από τις λογικές συμβάσεις έχει μειωθεί πάρα πολύ. Τα τελευταία δεδομένα που έχουμε από το 2012, τα οποία δημοσιεύτηκαν 2013-2014, μιλάνε για 61% πλέον μονοκάλυψη. Δηλαδή 7 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο σε σχέση με το ποσοστό κάλυψης που είχαμε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Θα πρέπει όμως να προσεγγίσουμε το πόρισμα αυτό και με όλες αυτές τις αναλύσεις που προτείνουμε στη μελέτη μας, να το δούμε δηλαδή από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το πιο σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι χώρες εκείνες που έχουν ποσοστό κάλυψης από τη συλλογική σύμβαση κάτω του 40% διπλασιάστηκαν από το τέλος της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα. Στο δεξί τμήμα λοιπόν του πίνακα βλέπετε τις χώρες εκείνες που έχουν υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις, οι οποίες διατηρούν σταθερά τελικά ποσοστά. Στα αριστερά του πίνακα βλέπουμε τις χώρες εκείνες που έχουν σταθερό ποσοστό κάλυψης και παραμένουν πάνω κάτω ίδιες. Στο μέσο όμως του πίνακα βλέπουμε τις ε, χώρες εκείνες που κυμαίνονται από το 20 μέχρι το 60% χώρες στις οποίες μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σημαντική μείωση, διάβρωση αν θέλετε, της κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων. Εν τέλει, το 1 τρίτο του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττεται από το φαινόμενο αυτό. Δεν καλύπτονται δηλαδή εργαζόμενοι πλέον το 1 τρίτο αυτών από τις συλλογικές αυτές συμβάσεις. Ένα στου δέκα θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγω λοιπόν, ολοκληρώνω με το συμπέρασμα αυτό και οι συναδελφοί μου μπορούν να σα δώσουν και πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία το ποσοστό κάλυψη ήταν περίπου 70% στα τέλη τη δεκαετία του 90. Είχε παρουσιάσει στην αρχή τη δεκαετία του 2000 αύξηση και τώρα έχει φτάσει μόνο το 30-35%. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια δραματική μείωση, αλλά αντίστοιχα ποσοστά έχουμε δει και στην Ελλάδα και εν μέρει και στην Πορτογαλία. Θα έλεγα ότι ε, αυτό είναι και το πιο εντυπωσιακό πόρισμα, το οποίο το βλέπετε με διαφορετικά χρώματα εδώ πέρα και στους χάρτες που βλέπετε, πώς έχει διαμορφωθεί και πώς έχει μειωθεί τελικά η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνω και είμαι στη διαθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα κυρία Μαρία Νταπάσκα Μοσλήμα για το θέμα της επιρροής στην Πορτογαλία και πώς επέδρεσαν για 10 λεπτά παρακαλώ. Το λόγο. Ε, Καλημέρα σας. Ε, καλό μεσημέρι, μα σε όλους. Ο τίτλος της παρουσίασής μου είναι «Η επιρροή της Τρόικα στη διάβρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Πορτογαλία, αλλαγή των κανόνων και αποτελέσματα». Η αφετηρία, που δεν θα έχουμε βέβαια χρόνο να συζητήσουμε εδώ, ούτε και είναι στόχος, είναι πολύ σημαντικό για να δείξουμε και να καταδείξουμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Πορτογαλία από το 2011 και εντεύθυν το 12, και 14 και ένα τμήμα και το 15. Οι πολιτικές αυτές λοιπόν ήταν αποτέλεσμα σε εφαρμογή του μνημονίου στην Πορτογαλία η Τρόικα, κατά την άποψή μου, εκπροσωπούσε ένα επίπεδο ε, επεμβατισμού και παρεμβατισμού από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς που ε, προηγουμένως δεν ήταν αρμοδιότητα ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του Διεθνούς ε, Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή ενώ ανάμειξη στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στον καθορισμό των μισθών κλπ. Οπότε... Situation. Uh, ε, the memorandum of... Είναι έκτακτες περιστάσεις δηλαδή. Οι σοσιαλιστές το υπέγραψαν ε, στην προσωρινή κυβέρνηση ε, αυτό το πάγωμα των μισθών και κλείθη να το εφαρμόσει η συντηρητική κυβέρνηση. Και αυτός ο κυβερνητικό συνασπισμός δεν εφήρμοσε μόνο το μνημόνιο το τροικανό, αλλά ε, ε, πήγε και ακόμα παραπέρα σε ορισμένε περιπτώσεις, ε, έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν κάποια βασικά στοιχεία της εφαρμογή του μνημονίου, να δούμε τι αντίκτυπο είχε και να μας προβληματίσει και να σκεφτούμε που οδηγούν όλα αυτά. Λοιπόν, Κάτι που φάνηκε από την αρχή στο μνημόνιο ήταν αυτό το πάγωμα των μισθών και των ε, προαγωγών στο δημόσιο. Αυτό αυτόματα μπλόκαρε οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευση συλλογική για τέτοια θέματα στο δημόσιο τομέα παγώσαν οι μισθοί του δημοσίου από το 2011 μέχρι το 2015. time, uh, Ταυτόχρονα υπήρξε και ένα αίτημα να παγώσει ο uh, υποχρεωτικός ε, δεσμευτικός κατώτατος μισθός και αυτό είχε επιπτώσεις χρόνια ολόκληρα. Όχι μόνο στο εισόδημα ε, ενό σημαντικού τμήματος του εργαζόμενου πληθυσμού, αλλά είχε επιρροή και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Σε κάποιες ε, περιπτώσεις και σε πολλές, ε, ο μισθός που καταβάλλεται είναι ο κατώτατος. Όταν παγώνεις τον κατώτατο μισθό, ε, παγώνεις και μπλοκάρεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται με βάση τον καθορισμό του μισθού αυτού. Τι άλλαξε λοιπόν, άλλαξε το νομικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και ποιες ήταν οι βασικές διαφορές. Ένας από τους στόχους ήταν η αποκέντρωση. Η αποκέντρωση ε, κατά το μνημόνιο σήμαινε ευελιξία και ανταγωνιστικότητα των μισθών. Τι αποκέντρωση ήταν αυτή. Ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο 2008. Ήδη από το 2008 και ε, ο νόμος ε, εργατικός του 2009 όριζε ότι κανένα συνδικάτο και καμιά αντιπροσωπευτική δομή δεν θα μπορούσε να κάνει επιχειρησιακές συμβάσεις. Ε, και ήταν καινούριο αυτό. Ακόμα και αν είχαν την εντολή. Μέχρι το 2008 μπορούσαν να διαπραγματεύονται τις συλλογικές συμβάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε κάθε εταιρεία δηλαδή, όχι συλλογικές, ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρεία. Τώρα άλλαξε αυτό και σου λέει θα γίνεται μόνο εφόσον έχεις εντολή του συνδικάτου σου και σε εταιρεία που απασχολεί πάνω από 500 άτομα. Η Τρόικα ε, μείωσε το κατόφλι αυτό και ε, ε, πρότεινε, απέτησε βασικά, εκπρόσωποι μη συνδικαλιστές να μπορούν να διαπραγματεύονται με την επιχείρηση χωρίς εντολή του συνδικάτου. Τι έγινε λοιπόν στην εφαρμογή και μπορείτε να το δείτε εδώ με κόκκινο. Αυτή η ιδέα των διαπραγματεύσεων χωρίς εντολή από το συνδικάτο δεν εφαρμόστηκε διότι είναι αντισυνταγματικό αυτό στην Πορτογαλία. Ελήφθησαν όμως άλλα μέτρα όπως είναι οι μειώσεις των μισθών ή μάλλον οι μειώσει ε, του, αριθμού των εργαζομένων εταιρεία για να γίνεται αποκεντρωμένη διαπραγμάτευση και όχι κεντρική συλλογική. Αυτό είναι λίγο περίεργο στην Πορτογαλία και πρέπει να τα πω λίγο γρήγορα. Αν δείτε πόσα έχει η πυκνότητα των συνδικάτων στην Πορτογαλία, σύμφωνα με ένα Ινστιτούτο του Άμστερνταμ, είναι 18,5% οι εγγραμμένοι στα συνδικάτα. Αν δείτε όμως ποιες είναι οι εταιρείε και πώς είναι οι αντιπροσωπευτικές δομές, η Πορτογαλία βρίσκεται ως η κατεξοχήν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το επίπεδο, με το χαμηλότερο επίπεδο των εταιριών που έχουν κάποια συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Μόλις το 8% των εταιριών είναι αυτό. Και ποια ήταν η ιδέα της αποκέντρωσης εδώ. Μαζί με αυτό λοιπόν και τμήμα αυτού ήταν η αλλαγή που ζήτησε η Τρόικα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Μέχρι τότε ήταν αυτόματη αυτή η διαδικασία σχεδόν. Αρκεί να ζητούσαν οι κοινωνικοί εταίροι παράταση των συλλογικών συμβάσεων και αυτό γινόταν αυτόματα. Και μπήκε ένας νέος κανόνας ότι θα πρέπει να εκπροσωπούν το 50% των εργαζομένων αυτοί που διαπραγματεύονται και κάνουν τις συνεννοήσεις για να ζητήσουν να παραταθεί η διάρκεια της ε, συλλογικής σύμβασης. Αυτό ε, λειτουργήσε τρία χρόνια με δραματικά αποτελέσματα, όπως θα δείτε ολέθρια, και άλλαξε στο τελευταίο τρίμηνο του 2013. 14, συγγνώμη, για να υπάρξει κάποιος χώρος για παράταση, αλλά όχι τόσο αυτόματο ούτε να λύνει το πρόβλημα. Ένα τελευταίο που έχει όμως τη σημασία του είναι η ιδέα να μειωθεί η περίοδος ε, μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων. Και αυτό άλλαξε το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Επίσης υπάρχουν δυνατότητες τώρα ατομικών συμβάσεων, ε, διαπραγματεύσεων γύρω από το ωράριο χωρί να συμμετέχουν ούτε να εμπλέκονται καθόλου τα συνδικάτα. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι επίσης κάτι που στρέφεται κατά των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Προηγουμένως είπα ότι η κυβέρνηση ε, ενέκρινε κάποια μέτρα πέραν του μνημονίου. Ε, επέδειξε εκεί έναν υπερβάλλοντα ζήλο. Στο δημόσιο τομέα δεν πάγουσαν απλώ οι μισθοί, αλλά είχαμε και ονομαστικές περικοπές μισθών που ξεκίνησαν ήδη από το 2011 πριν από την Τρόικα και συνεχίστηκαν και όλοι οι μισθοί πάνω από 1.500 ευρώ υπέστησαν ονομαστικές περικοπές. Έκοψαν δώρα ε, Χριστουγέννων, διακοπών. Ε, από τις 35 ώρες που είχαμε στο δημόσιο τομέα πέρασαν στις 40. Ε, μείωσαν τις διακοπές και τις επίσημες αργίες και γενικώ εμπλόκαραν τις συλλογικές συμβάσεις στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό. Αντίστοιχα μέτρα ελήφθησαν σε σχέση με το πώς πληρώνονται οι υπερορίες και τέτοια πράγματα και διακοπές. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος τώρα των μεταρρυθμίσεων. Προχωρούμε. Σε ό,τι αφορά. Έχετε εδώ αυτό το πίνακα, θα μπορείτε να το μελετήσετε στη συνέχεια. Ε, τι συνέβη, βασικά να σας εξηγήσω τι έγινε. Ο συνάδελφος από το Eurofound εξήγησε πώς γίνονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και πώς, ποια είναι η κάλυψη. Υπό την έννοια το πόσοι συμμετέχουν, ενώ εδώ είναι δυναμικό. Τι γινόταν κάθε χρόνο, ποιες ήταν οι ροές, ποιες ήταν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, που ε, κατέληγαν και ποιος ε, και πόσοι εργαζόμενοι καλύπτοντο κάθε χρόνο, πόσες συλλογικές συμβάσεις είχαν υπογραφεί κτλ. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ και τι είναι σαφές, ότι υπήρξε σαφής μείωση των κλαδικών συμβάσεων, ενώ οι επιχειρησιακές συμβάσεις είχαν μια ελαφρά διακύμανση. Ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου από τις συλλογικές συμβάσεις, με ανανέωση των συμβάσεων ή με νέες συμβάσεις, μειώθηκε δραματικά από ένα εκατομμύριο και μάλλον χιλιάδες σε 400.000. Χάθηκε ένα εκατομμύριο και μετά 200.000 από το 2013 και μετά. Εάν δούμε ε, την κάλυψη αυτή, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δραματική το 2009 και 2010 και 2011 περίπου το μισό, το, οι μισοί εργαζόμενοι ε, καλύπτοντο από τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ. Δηλαδή μισή εργαζόμενοι. Ε, το 9. Ενώ το 12, 13 και 14 πέφτει δραματικά. Ποιε είναι οι τάσει τώρα εξέλιξη των μισθών. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια από το 2012 και μετά είναι πολύ μικρό εκείνο το κομμάτι του εργαζόμενου πληθυσμού που πληρώνονται σύμφωνα με τις συλλογικέ συμβάσεις και όσα αυτά, αυτές ορίζουν για τους μισθούς. Συνέπεια, μειώθηκε αισθητά ε, το εισόδημα από την εργασία στην Πορτογαλία. Και αν δείτε και άλλες ε, μελέτες και άλλα στοιχεία θα καταλάβετε ότι αυτό οδήγησε και σε ανισότητες και σε αύξηση της φτώχειας. Συμπέρασμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μέτρα που ε, αφορούν αυτή την αποκέντρωση, ακόμα και αν έχετε νέους νόμους και νέους κανόνες, δεν επηρέασαν καθόλου. Το πάγωμα ε, του κατώτου του μισθού και πιο αυστηρά ε, κριτήρια για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων είχαν σημαντική αρνητική επίπτωση. Νέοι ε, ε, κανόνες για τη λήξη και τη μετενέργεια επίσης είχαν πρόβλημα γιατί πολλές φορές ζητούσαν οι εργοδότες να τερματιστεί η ισχύ των συλλογικών συμβάσεων και υπήρχαν και άλλα μέτρα που δεν έλεγε το μνημόνιο, που αφορούσαν τις υπερορίες, τα επιδόματα, τα δώρα και τις διακοπές, που είχαν επίσης ανητικές συνέπειες. Τώρα στον ιδιωτικό τομέα οι ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις είχαν μπλοκαριστεί και ιδιαίτερα τα μέτρα που δεν προέβλεπε το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, που δεν ήταν μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας για τη μείωση και τον περιορισμό του κόστους ε, της εργασίας. Τι γίνεται τώρα μετά την Τρόικα. Δώστε μου ένα λεπτάκι παρακαλώ. Μόλις βγήκαμε από το μνημόνιο. Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Αύξηση του κατώτατου μισθού, πολύ μικρή μεν, πλην αύξηση. Από τα 400 85 ευρώ έγινε 505 και κάποιες αλλαγές στις ε, διαδικασίες επέκτασης και παράτασης. Υπήρξε κάποια μικρή αλλαγή, αλλά πολύ περιορισμένη. Το σημαντικότερο τώρα που έχουμε να, να πούμε και να σημειώσουμε είναι ότι υπάρχει ένας νέος πολιτικός κύκλος ε, με τη νέα κυβέρνηση, τη σοσιαλιστική με την υποστήριξη των Ιστερών κομμάτων από τον Νοέμβριο του 2015 για να γυρίσει η σελίδα της λιτότητας. Ήδη έχουν ε, λάβει κάποια μέτρα σημαντικά όπως είναι η σταδιακή κατάργηση των ε, ονομαστικών περικοπών, ε, επιστροφή στα 35 ώρες στο δημόσιο τομέα και η σταδιακή αύξηση του υποχρεωτικού και κατώτατου μισθού. Ταυτόχρονα η σοσιαλιστική κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα που δείχνει προσιλωμένη να προωθήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και το ωράριο, να καλύπτεται ε, σχεδόν όλο το φάσμα, να ε, προωθείται ο κοινωνικός διάλογος και γίνεται μια συνεχή συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποια μέτρα όπως είναι η, ισχύς, η διάρκεια της ισχύω των συλλογικών συμβάσεων ή μετενέργεια ή διαδικασίες παράτασης τους. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς θα αλλάξουμε τους κανόνες αυτούς ε, και τι θα ισχύει για τις συλλογικές συμβάσεις, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να επιστρέψουμε στην πρώτερη κατάσταση μετά από τον όλεθρο που μας έφερε το μνημόνιο. Ευχαριστώ. Και τώρα. σα ευχαριστώ. Η κυρία, η δόκτωρ Αουρόρα Τρίφ, κατάσταση στην Ρουμανία και σας παρακαλώ να περιορίσετε στα 10 λεπτά για να μην ε, μας αγριέψουν και οι διερμηνείς. Πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη 12.30. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να συζητήσω για τις συνέπειες ε, στις συλλογικές συμβάσεις των προγραμμάτων της Τρόικα στη Ρουμανία. Ε, αυτό που έχω να σημειώσω εγώ είναι ότι οδήγησε σε μία ριζική αλλαγή στις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις Τρόικα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στις εξής πτυχές. Πρώτον, τα μέτρα λιτότητας και οι συνέπειές τους στι ε, συλλογικέ συμβάσει. δεύτερον συνέπειε για τους εργαζομένου και του κοινωνικού εταίρου. και τρίτον πώς μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Και άμα κοιτάξετε, στην ε, ανάπτυξη σε σχέση ε, του ΑΕΠ στην ε, Ρουμανία. Όταν ήρθαν οι αλλαγές, η κυβέρνηση χρειάστηκε να, να δανειστεί χρήματα από την Τρόικα. Πάω στην επόμενη διαφάνεια και βλέπουμε ότι η Ρουμανία δανείστηκε 20 περίπου δισεκατομμύρια από την Τρόικα. Πολύ λιγότερα από ότι η Ιρλανδία, η Ελλάδα και άλλες χώρες. Παρ' αυτά όμως, η κεντροδεξιά κυβέρνηση της ε, Ιρλανδίας ε, εφάρμοσε κάποια από τα πιο ε, ριζικά μέτρα της Τρόικας και να κοιτάξετε επί της ουσίας στην προηγούμενη παρακαλώ διαφάνεια μιλήσαμε για τις συνέπειες για τους μισθούς στην Πορτογαλία. Είχαμε 25% περικοπές μισθών στην Ρουμανία και πέραν αυτού και πολλά άλλα επιδόματα περικόπηκαν ή χρειάστηκε ή υποχρεώθηκαν οι εργαζόμενοι να πάρουν υποχρεωτικά άδεια ε, κατά 10-20 μέρες, 10 ε, μέρες μερες κατα το οποίο οδήγησε σε περιορισμό των εσόδων τους από τους μισθούς κατά 20% και εδώ βλέπουμε μια διαρκή επιδείνωση από το 2012. Στο δεύτερο σημείο, στα τυπικά μέτρα, στα διαδικαστικά. Αυτά έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και αυτή είναι η κύρια συνέπεια του προγράμματος της Τρόικα. Οδηγεί δηλαδή στην απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Και στην επόμενη διαφάνεια που δείχνει την ενεργεία, η ενεργεία και η δισκαμψία στην αγορά εργασίας δεν υπήρχαν στην Ρουμανία. 7 και, μέχρι, 7 και 8, μεταξύ 7 και 8% των Ρουμάνων είχαν εγκαταλείψει τη χώρα από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ήταν ίσως ο λόγος, άμα δούμε στην επόμενη διαφάνεια θα ε, δείτε τα στοιχεία. Και στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τις κύριες αλλαγές στα ατομικά δικαιώματα που προκύπτουν. Είδαμε δηλαδή ότι είχαν περισσότερα δικαιώματα ή ε, εργοδότες ως προς την πρόσληψη και την απόλυση εργαζομένων και μάλιστα ακόμη και ε, συνδικαλιστών σε εταιρικό επίπεδο καθένας κατάσταση, δηλαδή πολύ πιο εύκολο να απολύονται συνδικαλιστές, η εισαγωγή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, χρόνου απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες του εργοδότη και κατέστη πιο εύκολο για τον, ε, ο εργοδότης να αλλάξει το φόρτο εργασίας για τον εργαζόμενο πριν προβλεπόταν πώς θα πρέπει να το διαπραγματευτεί με το συνδικάτο. Αλλαγές λοιπόν στα συλλογικά δικαιώματα, σε εθνικό επίπεδο, ε, λεγόμενος κοινωνικός διάλογος ε, του 2011, ο οποίος πραγματικά δεν είχε ε, καμία μορφή διαλόγου, δεν ελήφθησαν υπόψη από την κυβέρνηση των ΕΣΥΓΑ για τα νέα μέτρα κάρτης ή οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπορούν ε, να κάνουν διατομεακές ε, συμβάσεις, να κάνουν διαπραγματεύσεις διατομεακές, εθνικές συλλογικές συμβάσεις δηλαδή, δεν μπορούν να κάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Σε επίπεδο εταιρικό δεν υπήρξε καμία νέα συλλογική σύμβαση στον ιδιωτικό τομέα ως συνέπεια αυτής της απόφασης και όπως βλέπετε έχουμε μείωση από 21, το από τομεακές σε 7 μόνο τομεακές συλλογικές συμβάσεις, σε ε, κλαδικές συμβάσεις, στις οποίες ε, ε, έλαβαν μέρος οι εργαζόμενοι. Συλλογικές συμβάσεις λοιπόν υπάρχουν σε ένα βαθμό μόνο σε επίπεδο εταιρικό, αλλά και πάλι είναι πολύ πιο δύσκολη η διαπραγμάτευση και ιδίω καθίσατε διαπραγμάτευση δύσκολη με την αλλαγή του ορίου εκπροσώπησης των σωματείων για το, στο 50% από το 30% που οριζόταν παλαιότερα, όπως ακούστηκε και στην πρώτη παρουσίαση, είδαμε μαζική μείωση της δύναμης των συλλογικών συμβάσεων για τους πάντες μετά το 2010. Έπεσε στο 30% το 2014. Εδώ βλέπετε τον αριθμό των συλλογικών συμβάσεων σε κλαδικό επίπεδο που, εκπροσ... που διαπραγματεύτηκαν αντιπροσωπευτικές ε, συνδικαλιστικές ενώσεις. Έχουμε 15% μόνο συλλογικών συμβάσεων που έχουν διαπραγματευτεί τα σωματεία. Σε ορισμένε περιπτώσεις, όπως συμβαίνει δηλαδή και στην Πορτογαλία και την ε, Ελλάδα, ε, δεν διαπραγματεύτηκαν οι συνδικαλιστές αλλά οι εργαζόμενοι μόνοι τους τις συλλογικέ συμβάσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν ήταν, και ότι δεν ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα αυτό που προέκυψε ως συλλογική σύμβαση. Επίσης υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό 15% 4-5 και οι οποίες ε, διαλέχθηκαν με συνδικαλιστικά σωματεία για τις λογικές αυτές τις συμβάσεις και στην επόμενη διαφάνεια έτσι βλέπουμε τις πρώτες τέσσερις περιπτώσεις κλαδικά όπου βλέπουμε σε κλαδικό επίπεδο μεγαλύτερη ισχύ των σωματείων και καλύτερη σχέση τους με τους εργοδότες. Εδώ λοιπόν μας λένε τα σωματεία ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η διαπραγμάτευση για τη συλλογική ε, σύμβαση. Ωστόσο, Ε, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για συνδιαλλαγή, στην επόμενη περίπτωση βλέπουμε ότι υπήρξε μείωση του χρόνου εργασίας από 5 σε 4 μέρες για την θερινή περίοδο, άρα αντίστοιχα μειώθηκαν και οι μισθοί, ή μειώθηκε το εργατικό δυναμικό σε, μια, σε έναν κλάδο κατά 40%, ή ε, δόθηκαν μόνο συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τους νέους απασχολούμενους και αυτές ήταν οι καλύτερες περιπτώσεις. Και θα μείνω σε αυτή τη διαφάνεια για να πω το εξής στην τελευταία ε, εταιρεία Food 4, Food 4 που βλέπετε στον πίνακα. Δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση, άλλαξε κατά την ύφεση η ιδιοκτησία και η νέα διοίκηση είχε μια πολύ αυταρχική συμπεριφορά, η οποία συμπεριφορά οδήγησε τους εργαζόμενους στην απόφαση να φτιάξουν συνδικάτο, γιατί με αυτό δεν υπήρχε όπως έλεγα. Και τι κάνουμε λοιπόν εδώ σε σχέση με τις συνέπειες αυτών των αλλαγών στην νομοθεσία για τους εργαζομένους πάνω απ' όλα ε, ανεξαρτήτως εταιριών, επηρεάζονται ιδιαίτερα. Ο εργοδότης έχει πολύ περισσότερες εξουσίες και σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί η υλοποίηση των αλλαγών αυτών από την ισχύ των συνδικάτων, τη σχετική ισχύ του κάθε συνδικάτου, δηλαδή, συνδικάτου, δηλαδή το πώς, πόσους ή πόσο ποσοστό από τους εργαζομένους έχει ένα συνδικάτο σε μια εταιρεία. Ε, έχω περίπτωση συνδικαλιστή που μου λέει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρεία του είναι μέλη του συνδικάτου, αλλά δεν κινητοποιούνται, δεν δραστηριοποιούνται όταν έρθει η ώρα. οι μεταρρυθμίσεις έχουν σαν συνέπεια την, ε, τον όλο και μεγαλύτερο κατακαιρματισμό και τους διχασμούς μεταξύ των εργαζομένων, διαφοροποιήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει μονομερός ακόμη μέτρα. Αυτό αφορά και, την κεντροδεξι... και τον κεντροδεξιό και τον κεντροαριστερό συνασπισμό που ήταν στην εξουσία στο 2015. Μέχρι τώρα λοιπόν τι έχει γίνει για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Δύο τύποι πρωτοβουλειών σημαντική η μία της κέντρο αριστερής κυβέρνησης που ανέλαβε το 2012 την εξουσία με ένα πρωτόκολλο συνεννόησης με τη μεγαλύτερη οργάνωση εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, στο οποίο οριζόταν ότι θα ακολουθούνταν οι συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αλλά όπως βλέπετε εδώ από τις παρατηρήσεις της Τρόικα εδόθη η υπόδειξη να μην ακολουθηθούν αυτές, το βλέπετε στην παράθεση στο κείμενό μας. Δεν υπάρχει, λέει, ανάγκη για αναθεώρηση νομοθεσίας προκειμένου να προσαρμοστεί αυτή στις ε, βασικές ε, συμβάσεις των, του οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι και η οργάνωση και η κινητοποίηση των εργαζομένων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονό ότι μετά το 2009 άρχισαν να οργανώνουν σε πολυεθνικέ το χώρο ιδιαίτερα τη λιανική πώληση, τη πληροφορική. Η ε, ε, τα συνδικάτα και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Δάτσο, που έχουμε ένα από τα καλύτερα συνδικάτα αλλά βέβαια και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης ε, μπόρεσαν να εξασφαλίσουν αύξηση των μισθών άνω του 10% ε, το τελευταίο διάστημα, αλλά μόνο ύστερα από μια 16ημερη απεργία. Στα τελευταία μου σημεία, στις τελευταίες παρατηρήσεις, ελπίζω να σας έπεισα πως έγινε μια ριζική αποκεντροποίηση και μαζική ε, μείωση των ε, συλλογικών συμβάσεων και της καλύψής τους λόγω τη παρέμβαση τη Τροϊκά, Αυτό οδήγησε σε επιδείνωση συνθηκών απασχόληση και κατακαιρματισμό και ε, διχασμό μόνο των κοινωνικών εταίρων, ε, υποβάθμιση των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων ήταν η συνέπεια όλου αυτού και μια πρόταση για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διαφυλάξουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Ρουμανία θα έλεγα ότι αντίστοιχα με αυτό που λένε και οι κοινωνικοί εταίροι για να υπάρξουν συλλογικές, συμβα... πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία στην κατεύθυνση των βασικών συμβάσεων του Οργανισμού, του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα νομιμοποίησης για να ενισχυθεί η νομιμοποίηση. Γιατί ήδη κάποιοι ηγέτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το έλλειμμα νομιμοποίησης ε, συνδικαλιστές εργοποιούνται, αλλά ταυτόχρονα και εκπρόσωποι των εργοποιητών με τους οποίους μίλησα φαίνονται διατεθειμένοι να δεχθούν ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μας λένε όμως πάνω απ' όλα ότι χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη για τα δέτα συνδικάτα τα οποία έχουν μπορέσει να οργανώσουν συλλογικές διαπραγματεύσεις κτλ. Συνήθως έχουν την υποστήριξη αλλοδαπών συνδικάτων από τη Γερμανία και άλλες χώρες, παραδείγματι. Άρα μας ζητούν υποστήριξη και μας ζητούν επίσης ή δυνατόν Οικονομική υποστήριξη. Τελευταία ε, διαφάνεια για να σας πω ευχαριστώ και ότι βεβαίως περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να ομολογήσω ότι σαν πρώτο και ενδιάμεσο σχόλιο οφείλω να διαπιστώσω ότι δεν μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτηση, πρέπει να διακόψουμε. Θα συνεχίσουμε στις 3.30 ε, με τις επόμενες δύο παρατηρήσεις. Πάντως είναι πολύ σημαντικό για μένα να επισημάνουμε ότι η Τρόικα αν περνούσε το δικό της θα ε, επέβαλε την ε, ολοκλήρωση την υπογραφή της σύναψης συλλογικών συμβάσεων με συμμετοχή των σωματείων των συνδικαλιστικών μόνο στις 29 Φεβρουαρίου ε, και μεταξύ ώρας 12 και 0 πρωινής ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η εικόνα την οποία βλέπουμε και για την Ελλάδα και για την Ρουμανία. Μεταξύ του 2011 και του 2015 που ξέρω εγώ τη μελέτη που αφορά την Ελλάδα από τις 1.100 ε, συλλογικές συμβάσεις το 70% δεν έγινε με εκπροσώπηση συνδικαλιστικών σωματείων. Αυτό λέει η γερμανική έκθεση και από αυτές το, 80, ε, το 98% οδηγούν σε μείωση των μισθών. Αυτή είναι η εικόνα. Μέσα σε δύο χρόνια η κατάσταση επιδεινώνεται σοβαρά σε κοινωνικό επίπεδο, σε μισθολογικό επίπεδο στα κράτη στα οποία έχει ε, δραστηριοποιηθεί η Τρόικα. Και αυτά τα οποία ονομάζονται κράτη πληττόμενα από την κρίση του ΣΥΠΗΝ. Αυτό πρέπει να το διαπιστώσουμε και να έχουμε συνείδηση αυτής της εξέλιξης. Όπως είπα θα εμβαθύνουμε στη συνέχεια στην απογευματινή μας συνεδρία. Σας εύχομαι τώρα καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε στις 3.30 και πάει στην διάθεση.